Mes Σας προτείνω να αρχίσουμε τις εργασίες μας της κοινή αυτής συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής μαζί με τον κύριο Πέτερ Σίμων και την Επιτροπή ΤΑΞ. Εάν δεν υπάρχουν ε, θέματα στη Μέσια διάταξη εγκρίνεται. Σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Προέδρου θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία δέκα πολιτικών συμβούλων του Σουηδικού Κοινοβουλίου είναι προσκαλεσμένοι του Γκούναρ Χέκμαρκ και τους ε, καλωσορίζουμε. Έχετε μπροστά σας το κατάλογο του γλωσσικού καθεστώτος και σας υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι γίνεται άμεση αναμετάδοση των εργασιών μας. Και όπως ξέρετε επίσης η συνεδριά της τάξη είναι ανοιχτές στο κοινό. Ε, δίνω τον ε, λόγο στον πρόεδρο Σάιμον. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αντικαταστήσω τον κύριο Γουαλτιέρη και θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Μοσκοβισή και ευχαριστώ τον Πρόεδρο ε, Λαμασούρ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μετά την 11η Ιανουαρίου και μετά την τελευταία Ολομέλεια. Σήμερα θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πακέτο φόρο που ενέκρινε η Επιτροπή στις 28 Ιανουαρίου. Ε, δημόσια καλωσόρισα αυτό το πακέτο όπως γνωρίζετε γιατί ασχολούμαστε με το ζήτημα της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. τα τέλη, κατά τα τέλη του 2015 εγκρίναμε μία έκθεση για τη διαφάνεια, συντονισμό και εναρμόνιση στον τομέα της εταιρικής χρηματο... Ε, ε, φορολόγησης. Με συγχωρείτε. Το πακέτο είναι ένα σημαντικό βήμα αλλά είναι η απαρχή της ιστορίας μας θα θέλαμε να ακούσουμε τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν υπό μορφή follow-up των συστάσεων της, ε, στις εκθέσεις ΕΚΟΝ και ΤΑΞΕ. Όπως γνωρίζετε, η ΕΚΟΝ έχει διορίσει τους δύο εισηγητές ο κύριος Ντάριος Ροζάτη για την τροποποίηση της οδηγίας για την διοικητική συνεργασία για την αυτόματη ανταλλαγή ε, πληροφοριών σε σχέση με τη φορολόγηση των πολυεθνικών και ο κύριος Μπαγιέ για την οδηγία καταπολέμησης της φοροαποφυγής που ε, ορίζει και εναρμονίζει εντάσσοντας ορισμένες συστάσεις του ΟΣΑ. Η Επιτροπή Οικονομικών και Οικονομικών Υποθέσεων προσπαθεί να εγκρίνει, να δώσει τελική μορφή στις εκθέσεις όπως εγκρίθηκαν στις 26 Απριλίου και στις 23, 23 ή 24 Μαΐου θα εγκρίνουμε την έκθεση καταπολέμησης της φοροαποφυγής. Θα εγκριθεί δε στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς προτίθεται το ε, Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν αυτά τα δύο μη νομοθετικά στοιχεία. Τις συστάσεις δηλαδή, τις ε, τάξ και τις, επικοι... και τις ανακοινώσεις για την εξωτερική στρατηγική στο... Ε, στα θέματα φορολόγησης. Θα θέλαμε λοιπόν να σας καλωσορίσουμε κύριε Επίτροπε και σας δίνουμε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι ενώπιον σας σήμερα. Είχαμε ειδωθεί κατά τα μέσα Ιανουαρίου και θα ήθελα να σας μιλήσω για τις προτεραιότητες για το 2016. Προβήκαμε σε μία ανταλλαγή απόψεων κατά τα μέσα Φεβρουαρίου με βάση το πακέτο αντιμετώπισης της φόρα και σήμερα θα επεκταθούμε σε αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε αυτή είναι η τρίτη μου παρέμβαση στο Κοινοβούλιο, διότι όπως ξέρετε γίνεται και η διακοινοβουλευτική ε, διάσκεψη. Η παρουσία μου σημαίνει ότι προσδίδω μεγάλη σημασία στον διάλογο μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας μιλήσω για τον νέο Γενικό ε, Διευθυντή, των Stephen Quest, ο οποίος είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής ε, της Γενικής μας Διεύθυνσης όπως ήδη ανέφερα στην Ολομέλεια και επαναλαμβάνω, αυτό το πακέτο αποτελεί μία πρόοδο καταπολέμησης της φοροαποφυγής. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα σε σχέση με την φοροαποφυγή. Γνωρίζουμε ότι αυτή η μάχη συνεχώς ανανεώνεται γιατί πάντα υπάρχουν αδυναμίες στο σύστημα προς εκμετάλλευση και όπως πολύ ε, καλά γνωρίζουμε η τεχνολογία όπως και η φαντασία έχουν όρια. Θα πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι από αυτούς που προβαίνουν σε απάτες και να σκεφτούμε εις βάθος τα ζητήματα για να νικήσουμε. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο ε, ζητήματα σε σχέση με την παρέμβασή μου τον Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Θα ήθελα καταρχήν να μπούμε στις λεπτομέρειες του κειμένου που ε, μελετήσατε μετά την έγκρισή του, καθώς και να σας ε, καταδείξω πώς το πακέτο ανταποκρίνεται στις συστάσεις των δύο επιτροπών που παρίστανται απόψε. Καταρχήν πώς ε, μπορούμε να ανταποκριθούμε με τα άμεσα μέτρα. Βεβαίως έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες γιατί θέλουμε να δώσουμε τέλος σε μια κατάσταση κατάφορης παραβίασης, δηλαδή εκεί όπου πολλές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι πολυεθνικές στην ουσία καταβάλουν πολύ χαμηλούς φόρους αντιπαρερχόμενες στη, ε, στα φορολογικά καθεστώτα. Και κατά συνέπεια οδηγούν στην αποδυνάμωση των φορολογικών αρχών και των, ε, του, του δημοσίου, των δημοσίων εσόδων, κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Για να απαντήσω σε αυτά τα ε, δεδομένα, το πακέτο το οποίο υπέβαλα βασίζεται σε τέσσερις ε, πυλώνες στην πραγματική θέση των επιχειρήσεων και όχι τη θεωρητική τους θέση, δηλαδή θα πρέπει να καταβάλουν ε, το φόρο με βάση τα κέρδη, επίσης μία φορολογική διαφάνεια, μία, ε, έναν ανταγωνισμό ο οποίος να είναι δίκαιος και διαφανής και καθώς, ε, καθώς και τη σωστή διάρθρωση της στάσης μας ως προς την ως προς την εξωτερική πολιτική και τον εξωτερικό πυλώνα. Νομίζω ότι στη, στην ουσία όταν μιλώ για το γεγονός ότι θα πρέπει να καταβάλλονται οι φόροι εκεί όπου υπάρχουν κέρδη, φαίνεται σαν να παραβιάζω μία πόρτα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Η πόρτα αυτή δυστυχώς είναι κλειστή, εκεί όπου δεν θα έπρεπε. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προβούμε σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Τα μέτρα που προβλέπονται από την οδηγία για την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής και της αποφυγής στοχοθετούν, βάζουν στο στόχαστρο συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι οποίες καταχρώνται τις θέσεις τους. Γι' αυτό έχουμε να κάνουμε με τρία φορολογικά στάδια έχουμε να κάνουμε με τις υβριδικές μορφές ή οντότητες, οι οποίες στην ουσία εκμεταλλεύονται τις φορολογικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ χωρών, επίσης τις ελεγχόμενες ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες στην ουσία εξάγουν τα κέρδη εκεί όπου φορολογούνται κατά πιο ε, πλεονεκτικό τρόπο. Επίσης υπάρχουν Υπάρχει και η μεταφορά στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων, εκεί όπου φορολογούνται χαμηλότερα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτά τα μέτρα τα βρίσκεται και στις δικές σας, στα δικά σας ψηφίσματα. Θέλουμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση αυτών των φορολογικών συμβάσεων ε, μιλάμε για το περίφημο σαλαντάζ φισκάλ, για το forum shopping και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα και με βάση τις συστάσεις του ΟΣΑ. Υπάρχουν ε, βεβαίως και θέματα δικαίου που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή μπορούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν τις διμερείς φορολογικές συμβάσεις έτσι ώστε να υπάρχει άλλη φορολογική βάση μεταξύ κρατών μελών. Και πολλοί θα επιθυμούσαν να μην ξεφύγουμε από θέματα εθνικής κυριαρχίας, να μην τα υπερβούμε δηλαδή δηλαδή να μην υπερβούμε το πλαίσιο της οδηγίας. Βεβαίως υπάρχει και το πολιτικό επίπεδο, διότι θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους στις προσπάθειές μας. Και φυσικά τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει τώρα να δώσουν μία απάντηση. Στα πλαίσια του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ είχαμε μία πολύ ε, καλή συνεργασία αλλά ορισμένα κράτη-μέλη επέμειναν υπέρ του γεγονότος ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε την πέψη, τα ΠΕΠΣ, γιατί έχουμε την εσωτερική μας αγορά και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δικές μας συμβάσεις. Αν δεν το κάνουμε, τότε δεν τηρούμε τη νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε το συνολικό πακέτο. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι η φορολογική διαφάνεια. Με βάση το, την εποπτεία και το reporting θέλουμε να υπάρξει φορολογική διαφάνεια. Ξέρετε ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της οδηγίας μετά από τη σύσταση του ΩΣΑ. Προβλέπουμε την άμεση και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών και το συζήτησα και με τον κύριο Ροζάτη, ο οποίος ε, ε, επεξεργάζεται αυτό το θέμα. Ξέρω ότι μερικοί από εσά θα ήθελαν να κινηθούμε περαιτέρω και να έχουμε δημόσιες δηλώσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, δημόσιο reporting δηλαδή. Αυτή είναι και η δική μου επιθυμία. Η Επιτροπή όμως θα ζητήσει την μεταφορά αυτών των δεδομένων μεταξύ φορολογικών αρχών και όπως ξέρετε γίνεται μια μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια τον Απρίλιο θα δημοσιεύσουμε τη θέση μας. Αυτή η πρόταση θα συνοδεύεται από τη μελέτη αντικτύπου μετά από μία δημόσια κροματική διαδικασία. Θα πρέπει ε, να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση μέσα στα πλαίσια της εξίσωσης αυτής και φυσικά να γίνει και μία δημόσια συζήτηση αναγνωρίζοντας και τα όρια μας. επεξεργαζόμαστε αυτό το σημείο, αλλά θα κινηθούμε σε δύο στάδια, γιατί μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια δικαίου, η νομική ασφάλεια, όπως προτάθηκε και από τον ΩΣΑ. Και βασιστήκαμε και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, ο τρίτος πυλώνας ορίζει τη θέσπιση ε, μιας, ενός φορολογικού ανταγωνισμού, ο οποίος να είναι δίκαιος και η μή οι ΜΜΕ καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις να την χάνουν τις ίδιες μεταχείρισεις. Πολλές ε, μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη δεσπόζουσα θέση τους για να ε, μην καταβάλουν φόρους ή να προβούν σε φοροαποφυγή. Θεωρούμε λοιπόν ότι πολλές φορές ο, ο φόρος που καταβάλλεται από τις ε, ΜΜΕ είναι κατά 30% υψηλότερος από αυτόν που καταβάλουν οι πολυεθνικές. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να είναι πιο επιθετική προς τις πολυεθνικές οι οποίες έχουν ε, τα, μέσα να φοροαποφύγουν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια, ένας δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών με ίδια φορολογική βάση. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το νέο πλαίσιο. Δυστυχώ δεν ισχύει παντού κάτι τέτοιο. Πρόκειται για μια άδικη κατάσταση όπου ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη κατά των καταχρήσεων δεν βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να, υπάρχει, να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και να τηρήσουμε και το εταιρικό πλαίσιο κατά δίκαιο τρόπο. Τελευταίος πυλώνας θέλουμε να ορίσουμε μια πραγματική εξωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση τις ε, πρωτοβουλίες μας πιστεύουμε ότι θα δώσουμε μια παγκόσμια απάντηση σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στην φόρο αποφυγή. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρεία συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών εταίρων, έτσι ώστε να προωθήσουμε την ε, χρηστή διεθνή φορολογική διακυβέρνηση. Και φυσικά θα αντιμετωπίσουμε και τα κράτη πιο επιθετικά, τα κράτη τα οποία δεν τηρούν τις προδιαγραφές, δηλαδή τις χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται και αυτό αφορά και συνεργασία με τρίτες χώρες μέσα στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού καταλόγου. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις νομικές αρχές. Ήδη η Επιτροπή μελετά αυτά τα κριτήρια τα οποία θα μπορέσουμε να υποβάλουμε φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα δυνατά στοιχεία από τις εθνικές νομοθεσίες και αυτό το ζήτημα θέλουμε να προωθήσουμε. Θα ήθελα τώρα να φτάσω σε ένα σημείο που χρειάζεται να συζητήσουμε για την ανταγωνιστικότητα και την ε, ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τα μέτρα που έχουμε μέσα στη δέσμη αυτή δεν είναι εχθρικά προς τις επιχειρήσεις του αντίον μάλιστα. Θα επιτρέψουν μια συντονισμένη προσέγγιση στο πρόβλημα της φοροαποφυγής και δεν θέλουμε ένα ε, μοσαϊκό εθνικών νομοθεσιών που θα παρέβλαπτε βέβαια την εσωτερική αγορά και άρα και την οικονομική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων γιατί ο κατακαιρματισμός και η νομική αβεβαιότητα κοστίζουν ακριβά. Τα μέτρα που προβλέπουμε θα έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση μιας, ενός φορολογικού συστήματος υπέρ των επιχειρήσεων που δρούν με βάση τους κανόνες και όχι αυτών που παίζουν με τους κανόνες. Και επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνη της σε αυτόν τον αγώνα κατά της φοροαποφυγής. Πάνω από 100 κράτη και ε, περιφέρειες και επικράτειες έχουν δεσμευθεί με, να ακολουθήσουν γρήγορα τις συστάσεις του ΩΣΑ στη διάσκεψη κορυφής του, του G20 στην Ατάλια τον τελευταίο Νοέμβριο και αυτό σημαίνει ένα πραγματικό κίνημα παγκόσμιο κατά του ε, επιθετικού φορολογικού προγραμματισμού. Πρέπει λοιπόν εμείς να παρακολουθήσουμε και να καθοδηγήσουμε αυτή την κατάσταση, αυτή την εξέλιξη. Για το Συμβούλιο, λοιπόν, ξέρετε, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσει. Έγινε το Συμβούλιο Κοφίν ε, τη προηγούμενη Παρασκευή που σα ανέφερα, ε, όπου συζητήθηκε καν και επί της ουσίας οι προτάσεις, αλλά και το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησή τους. Θα έχετε ε, από τις επαφές σας με την Ολλανδική Προεδρία, άλλωστε διαπιστώσει και επιβεβαιώθηκε και από την συνάντηση του ΕΚΟΦΗΝ, ότι η Προεδρία με το φίλο μου Γέρουν Ντάισελμπλουμ έχει ετοιμάσει ένα πολύ εντατικό και φιλόδοξο πρόγραμμα. Ο Υπουργό των Κάτω Χωρών θέλει να προωθήσει το ταχύτερο δυνατό τι εξελίξει και τι αποφάσει και εγώ τον εγκρίνω τι επιλογέ του, τον ενθαρρύνω σε αυτέ και τον ε, ακολουθώ. Και θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στον κίνδυνο της ε, ε, αποδιάστρωση αυτών των προτάσεων, καθώς ορισμένοι θα ήθελαν να περιορίσουν τη φιλοδοξία στην υιοθέτηση μόνο των στοιχείων BEPS του ΩΣΑ. Δεν θα θέλαμε να γίνει αυτό, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε σχέση με τα όσα ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να μεταφαρθούν αυτές οι συμφωνίες BEPS του ΩΣΑ. Είναι όρος επιτρονού κάνευ. Είναι το ελάχιστο απαραίτητο να υιοθετηθεί ε, αυτό το πακέτο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την φοροαποφυγή στην εσωτερική αγορά. Και κλείνοντα, ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα με πιο λεπτομερεί ε, τοποθετήσει, θα ήθελα να σημειώσω ότι στηριζόμαστε στην ελπίζουμε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου για του επόμενου μήνε για να διατηρηθεί αυτή η πολιτική επικαιρότητα και ορμή που υπάρχει στην παρακολούθηση των θεμάτων. Χωρίς εσάς το πακέτο αυτό δεν θα είχε προωθηθεί ασφαλώς. Τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στις εκθέσεις που παρουσιάστηκαν πέρυσι από τις δύο επιτροπές σας, ΕΚΟΝ και ΤΑΞΕ, δείχνουν ότι τα θεσμικά μας όργανα είναι ε, ήδη προσανατολισμένα προς την ε, αναγνώριση αναγκαιότητας υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού προγραμματισμού και την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας. Ξέρω ότι αναζητείτε τον προσδιορισμό των επόμενων βημάτων για τις συστάσεις της τάξης και της ΕΚΟΝ. Ξέρετε ότι είναι δεκάδες αυτές οι συστάσεις εγώ τώρα εισαγωγικά ανέφερα κάποια σημεία σύγκλησης, αλλά δεν είναι δυνατόν να εκθέσω κάθε λεπτομέρεια και κάθε μία από αυτές τις ε, συστάσεις σας για να ε, απαντήσω στην καθεμία χωριστά. Ωστόσο θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει την ε, πρότασή της ως ανταπόκριση στα κοινά ψηφίσματα τάξη και έκον. Ε, παίρνουμε πολύ στα σοβαρά αυτό το καθήκον και ελπίζουμε να μπορέσουμε να επανέλθουμε το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε σημείο χωριστά στις προτάσεις σας και στις δράσεις που θα έχουν αναλυφθεί σε σχέση με αυτές, ε, όπως είπα σε κάθε ένα από τα σημεία των ε, συστάσεων των ψηφισμάτων σας. Δέσμευσή μου είναι ε, η πολύ στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, θα συνεχίσει Άλλωστε έχουμε πολύ καλές σχέσεις και με τον πρόεδρο Σιμών και μπορεί να το επιβεβαιώσει και εκείνος ότι έχουμε ε, στρατευτεί στην ε, διαφάνεια σε σχέση με την πρόσβαση στα έγγραφα και οπότε που ανέλαβα εγώ καθήκοντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδείξει και επιδείξει διαφάνεια χωρίς προηγούμενο το λέω ξεκάθαρα και περίφραστα ότι έχουμε δώσει πρόσβαση στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα έγγραφα του κώδικα συμπεριφοράς ε, που έχει στη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ίδρυση, από την θέσπιση αυτού του κώδικα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί στο παρελθόν. Και ε, ένα νέο ένα κτίριο λάκτισμα εδόθη εχθές, ύστερα από τις ανακοινώσεις του Προέδρου Γιουνκέρ. Άπαξ και μα δοθεί και η απάντηση του Κοινοβουλίου ω προ τη διατυπώση των διαβουλεύσεων in camera και κλεισμένων των θηρών μέσα στι δικέ σα ε, αίθουσε συνεδριάσεων, ε, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε από κοινού τους απολογισμούς οποίους θα έχουμε ε, καταλήξει από τις συνεδριάσεις μας για τον κώδικα συμπεριφοράς όπως ακριβώς το ζητήσατε και εσείς κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι ε, κύριοι, κύριοι Πρόεδροι, ε, αυτά ήταν τα λίγα λόγια που ήθελα εισαγωγικά να σας ε, μεταφέρω. Είμαι στη σας για να δώσω κάθε λεπτομερή απάντηση για τις επιλογές που εκφράζονται μέσα από το πακέτο αυτό και για να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την συνοχή και την παρουσίαση του πολιτικού δρόμου από εδώ και μπρος ο πρόεδρος Λαμασού. Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Μοσκοβιστή, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερω για τη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας και της, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημών προσωπικός των υπηρεσιών σας, ε, της Επιτρόπου Φερστάγκερ και των δικών της υπηρεσιών που θα δούμε σύντομα, για την τελευταία σας παρατήρηση, την κοινοποίηση δηλαδή των εγγράφων. Ε, θα σας ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερος για την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας, των διαπραγματεύσεων και της ανταλλαγής των απόψεων που οδηγούν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όπως το έχουμε ζητήσει εξ αρχής, δηλαδή την επίλυση νομικών αλλά και πρακτικών προβλημάτων. Τα οποία θα συζητήσουμε εδώ, αλλά την επόμενη εβδομάδα με μια συντονιστική συνεδρίαση Tax ε, θα κοιτάξουμε αυτές τις διατυπώσεις να τις, να τις εκφράσουμε στο δυνατόν πιο ξεκάθαρα και πρακτικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Μοσκοβισή και τώρα παίρνουμε στη φάση ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα δίνουμε πεντά λεπτά σε κάθε περίπτωση που θα τηρούνται αυστηρά, πολύ αυστηρά. Ο κύριος Παύλος Σάλβα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ μεταξύ μας. Βεβαίως ε, συμμεριζόμαστε τους κοινού στόχους και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν αυτές οι δύο επιτροπές μετά από συντονισμό έχουν έχουν ενταχθεί στις δικές σας προτάσεις. Αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. Τα λυπηρά γεγονότα που γνωρίσαμε αποτελούν ευκαιρία για να προχωρήσουμε σε μία πιο δίκαιη φορολογική βάση της Ευρωζώνης, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να ε, φοροαποφεύγουν ή να αποδέχονται αυτή την φοροαποφυγή ε, ως προς χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της ε, εκπαίδευσης, της υγείας και ούτω καθεξής. Πολλά προσμένουμε να ακούσουμε από το Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής μας ε, κάνατε ορισμένες νήξεις, αλλά μέχρι πού νομίζετε το, το Συμβούλιο θα προχωρήσει προς την δίκαιη αυτή φορολόγηση. Ποια θα είναι η φιλοδοξία του Συμβουλίου. Επίσης, σε σχέση με τη ε, διεθνή συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα. Χρειάζεται μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία Πώς θεωρείτε ότι οι αρχές των ΙΠΑ είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν έτσι ώστε να υπάρξει δίκαιη φορολογική βάση και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ευχαριστώ. Καταρχήν για το Συμβούλιο και επανέρχομαι στις συζητήσεις του της προηγούμενης Παρασκευής στο ΕΚΟΦΗΝΟ εδώ και 15 θα έλεγα μήνες έχουμε καλές σχέσεις με το Συμβούλιο και ξέρετε ότι έχει προχωρήσει την υιοθέτηση των, από, των προτάσεων για τις ε, ε, φορολογικές προκαταρκτικές αποφάσεις, τα tax rulings. Μια πρώτη μου λοιπόν εντύπωση είναι θετική. Βλέπουμε ότι όλοι παρακολουθούν τους γενικούς στόχους, την πολιτική βούληση και για άλλη μια φορά χαιρετίζω την Ολλανδική Προεδρία η οποία αφήνει το ίχνος της και σημειώνει ότι πρόκειται για ε, απόλυτη προτεραιότητα και ότι θέλει να προχωρήσει γρήγορα στον εαυτό. Αλλά, αλλά με μια μικρή επιφύλαξη και προειδοποίηση, θα πω ότι μπορεί να φαίνονται καταρχήν ε, καλής, ε, κοινή λογική οι προτάσει, να ξεκινήσουμε με τα BEPS και μετά να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Σε αυτήν όμω την προσέγγιση ενδέχεται να χάσουμε την γενική ε, λύση, τη γενική προσέγγιση, η οποία θα σήμαινε και ρήγματα στο ε, πλέγμα το νομοθετικό που θα εισαγάγουμε. Κάτι το οποίο θα σήμαινε ότι θα αρχίσουμε να χάνουμε πόντους, να χάνει πόντους το πλεκτό αυτό, ή να διαλύεται το οικοδόμημα ε, πριν καλά-καλά οικοδομηθεί σωστά. Γι' αυτό είναι και η βούληση, η στεναρή βούληση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου ασφαλώς να πιέσουμε με τρόπο ώστε να προχωρούσαν πράγματα γρήγορα και με τρόπο ολοκληρωμένο. Είναι συνενετικά όσοι έχουν συζητηθεί και στο Συμβούλιο και στην G20 και βέβαια στην Επιτροπή οι συζητήσεις μας, τόσο συνενετικές που δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να παρεμποδίσει αυτές τις εξελίξεις, όσο και αν κάποια κράτη μπορεί να έχουν τη δική του το καθένα προσέγγιση. Ως προς τη διεθνή συνεργασία και τις ΗΠΑ, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, όχι δυστοκίες αλλά εν πάση περιπτώσει παρατηρήσεις ε, που άλλωστε γνωρίζετε και από τις τελευταίες επιστολές της Υπουργού των Εξωτερικών. Ωστόσο οι Αμερικανοί θα γνωρίζετε οπωσδήποτε και εσείς ήταν εκείνοι οι οποίοι πρώτοι εκκίνησαν την υπόθεση BEPS. Με τον Σαούλε, τον Νόσμπορν, τον Γκρίλι, τον Δεκίτος και βέβαια τον υποφαινόμενο που, θέσαμε ε, τα θεμέλια αυτή τη προσπάθεια. Θα συνεχιστούν άλλωστε οι εργασίε τη G20 που προβλέπεται την επόμενη εβδομάδα να συνέλθει σε επίπεδο των Υπουργών Οικονομικών ε, στη Σανγκάη, μάλλον οικονομία στη Σανγκάη ε, και έτσι καταλήγω στο συμπεράσμα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και όχι μόνο και οι κύριε χώρε του G20 ε, έχουν μπει σε έναν χώρο που δεν θα σταματήσει πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να μηδενιστεί το χρονόμετρο για να παρακολουθούμε το χρόνο μας. και να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι βέβαια πώς εξελίσσεται το χρόνος ομιλίας. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Ελίζα Φερίρα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Επίτροπο για την σημερινή του παρουσία και για όλη του την εργασία εδώ πρόκειται για μια κοινή συνεδρίαση δύο σημαντικών επιτροπών, της ΕΚΟΝ και της ειδική Επιτροπής ε, ΤΑΞ και σε αντίθεση με το παρελθόν ε, η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες δημοσιονομικού και φορολογικού χαρακτήρα. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω τις εξής ερωτήσεις. Στις επόμενες ε, εβδομάδες θα γίνουν συστάσεις αναχώρα στο φορολογικό τομέα, δηλαδή στο εθνικό φορολογικό πλαίσιο. Όμως, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ίσως ε, θα έπρεπε να ασχοληθείτε και με θέματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μακροοικονομικές ανισότητες, γιατί μιλάμε για δεδομένα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ΟΣΑ, θα γίνει σύγκριση στοιχείων και θα δούμε κατά πόσο υπάρχει απόκληση από τη φορολογική βάση, την θεμητή φορολογική βάση. Θα εισαχθεί και αυτό το στοιχείο στη δική σας προσέγγιση μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας. Δεύτερον, πότε θα γίνουν συστάσεις προς τις χώρες. Θα θέλαμε να υπάρχει προστασία της φορολογικής βάσης θα θέλαμε το Συμβούλιο να συνεργαστεί, να μην αποδυναμώσει τις προτάσεις, αλλά στην παράγραφο 172 προτείνουμε στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το άρθρο 116 των συνθήκων, έτσι ώστε να μην υπάρχει, ε, να μην πρέπει να ληφθούν αποφάσεις με ομοφωνία. Αυτές είναι οι τρεις ερωτήσεις που θα ήθελα να υποβάλω. Ευχαριστώ. αναχώρα. Ναι, συμφωνώ ως προς το ζήτημα της ε, φορολογίας και βέβαια το πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι η κάθε στην ε, πρακτική των επιθετικών ε, φορολογικών προγραμματισμών. Καταγράφεται ήδη και στην ανάλυση μας αναχώρα. Εμείς θα φωτίσουμε ιδιαίτερα αυτή τη διάσταση. Είναι νωρί, δεν μπορώ να δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες, γιατί εξορισμού είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί την επόμενη εβδομάδα από την Επιτροπή στη Συλλογική της Μορφή, ε, όπως άλλωστε θα εξεταστούν και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αυτή τη στρεβλωτική δηλαδή διάσταση, γιατί θέλουμε στο δυνατόν περισσότερη ε, αξιοπιστία σε σχέση με το θέμα των υπερβολικών ελλημάτων. Πρέπει να βρούμε δηλαδή το πλαίσιο των, ε, συγνώμη, των υπερβολικών πλεονασμάτων. Ένα υπερβολικό πλεόνασμα της ζώνης ευρώ που σημαίνει ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις χώρες που χρειάζονται περισσότερο η προσπάθεια αλλά και αυτές που έχουν μεγαλύτερο περιθώριο αλλά αυτές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια ακόμη και είναι πίσω να τύχουν περισσότερων επενδύσεων. Για το τωρινό πλαίσιο και το άρθρο 16 δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ σας λέγω. Ε, βεβαίως η Επιτροπή είναι πάντα έτοιμη να αξιοποιήσει κάθε ε, δυνατότητα αλλά παραδοσιακά θεωρούμε ότι οι φορολογικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε με ομοφωνία. Πολλές φορές με πολύ ε, μεγάλη δυσκολία και παρεμπόδιση των εξελίξεων λόγω της ομοφωνίας. Ωστόσο, είμαστε αισιόδοξοι γιατί είναι κάτι το οποίο τόσο πολύ ζητεί και η κοινή γνώμη και τόσο πολύ έχει προβληθεί και έχει ε, συζητηθεί που και οι κυβερνήσεις και τα κράτη θα ακολουθήσουν. Πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε με απόλυτα σαφή και επακριβή τρόπο, έτσι ώστε οποιοδήποτε προσπαθήσει να προβάλλει ψευδοτεχνικού χαρακτήρα ε, ε αντεπιχειρήματα να καταγγέλλεται και να μπορούμε να παρακολουθούμε τον φόρο φυγά ή τον φόρο αποφεύγοντα ε, επιχειρηματία. Επιχείρηση καλύτερα. Και πάντως, σε αυτή την προσπάθεια στηρίζομαι στη δική σας υποστήριξη. Για την προστασία της ε, φορολογίας σχέση με την νομοθεσία τη σχετική με τον περιορισμό των ε, δημοσίων δαπανών. Ναι, βεβαίως και αυτό μπορεί να μπει μέσα στη συζήτηση, ε, αλλά θα το δούμε, όπως είπα, στις συστάσεις μας που εξορισμού αφορούν την κάθε χώρα χωριστά. Ευχαριστώ όλοι ο κύριος Λαμασούρ. Τρέχει το χρονόμετρο. Ο κύριος Ashley Φόξ για, το, ε, για τους Ευρωπαίους Μεταρρυθμιστές. E ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Επίτροπο. Η ομάδα μου καλωσορίζει τις προτάσεις σας εκείνες που σκοπό έχουν να εφαρμόσουν τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν λεφθεί σε επίπεδο όσα σε ό,τι αφορά τη διάβρωση ε, της βάσης και τη μετατόπιση του κέρδους. Αυτές οι παρουσιάσεις, λοιπόν, αυτές οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο θα πρέπει να μεταφραστούν σε διεθνές επίπεδο και έχει κάποιο ρόλο να μεταγραμματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει συνοχή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συστάσεων αυτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά έχω ανησυχίες για το πακέτο σας που ξεπερνάει τις ε, συστάσεις BEPS του ΟΣΑ. Μπορώ να ρωτήσω για παράδειγμα γιατί προτείνεται ε, ρήτρα switch over και ένα exit tax, ένα φόρο εξόδου. Δεν προβλέφθηκε ούτε το ένα ούτε το άλλο από τις συστάσεις του ΟΣΑ και τα δύο μέτρα θεωρώ ότι θα ε, έχουν σκοπό να περιορίσουν την μετακίνηση των κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μάλλον παρεμποδίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν την ενθαρρύνει. Κατά δεύτερον, η πρόταση, η πρότασή σας για τα ευρυδικά είναι πολύ διαφορετική από αυτή που πρότεινε ο ΣΑ και είναι πιο χαλαρή όλος περίεργος. Γιατί, γιατί δεν ισχύει σε όλες τις διευθυντήσεις τρίτων χωρών παρά τη σαφή επιθυμία του ΩΣΑ να υπάρξει σύνοχη και συνέπεια σε διεθνές επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι πρόημο να συμπεριληφθούν ένας ε, νόμος ε, περιορισμού των τόκων, μιας και δεν έχει ολοκληρώσει τις σχετικές έρευνες και μελέτες η ομάδα του ΩΣΑ. Αν θέλουμε λοιπόν και απότατος στόχος μας είναι να υπάρχει συνοχή σε διεθνές επίπεδο, γιατί προκαταβάλλεται τις αποφάσεις του ΩΣΑ. Πού θα ακολουθήσει ο υπόλοιπο κόσμος, δεν θα βάλει αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ανταγωνιστικό, σε μια ανταγωνιστική μειονεκτική θέση, αν τελικά αποφανθεί διαφορετικά ο ΩΣΑ. Και τέλος, αποδέχεστε ότι χρειάζεται συντονισμένη παγκόσμια δράση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Και αν ναι, γιατί αγνοείτε τις συστάσεις του ΩΣΑ σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες άλλες ε, υπερβαίνετε ακόμα αυτές τις συστάσεις ή μήπω ακολουθείτε τη δική σας πολιτική ατζέντα για πιο πολύ Ευρώπη, όποιο και αν είναι το ερώτημα στο οποίο απαντάτε. Ευχαριστώ, ο κύριος Επιτροπός. Οπωσδήποτε θα απαντήσω ξεκάθαρα στο τελευταίο αυτό σημείο. Δεν υπάρχει πολιτική ατζέντα η επιδίωξη ούτε της Επιτροπή στο σύνολό τη, ούτε κάθε επιτρόπου χωριστά ή ουδήποτε επιτρόπου χωριστά ασφαλώς βάση των πάντων είναι οι εργασίες του ΩΣΑ όπως τις ε, ε, ενέκρινε το G20 στην Ατάλια. Η εφαρμογή όμως των BEPS, της διάπλωσης βάσης, προλογικής βάσης και μεταφοράς κερδών, δεν θα αρκέσει για τον εξωτό λόγο ότι αποτελούμε εσωτερική αγορά. Είμαστε λοιπόν εσωτερική αγορά και έχουμε ρυθμίσεις και νομολογία του δικαστηρίου που μπορεί να οδηγήσει, να οδηγήσουν σε δυνατότητες για περαιτέρω φόρο απάτη και φόρο αποφυγή και άρα είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε πέραν των BEPS. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα προχωρήσουμε και, ο λόγος για την ε, κατάθεση της πρότασης και των διατάξεων switchover που επιτρέπει στα κράτη να ε, βγουν από την ε, βάση αυτή της έδρας για τα κέρδη και επίσης η στρατηγική, εξωτερική στρατηγική που μιλάει για μια χρηστή φορολογική διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο και μια προσέγγιση κοινή για έναν κατάλογο μαύρη λίστα των κρατών που δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές και τις συμφωνίες η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στη τελευταία ανάλυση έχει οδηγήσει την νομοθεσία και έχουμε αναγκαστεί να προσαρμοστούμε σε αυτέ. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν περιοριστούμε στα BEPS, χωρί να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση οικονομική από την υπόλοιπη διεθνή ε, κοινότητα, τι κάνουμε, αφήνουμε στον φοροφυγά, στην ε, πολυεθνική, πεδίο για να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Προσπαθούμε ακριβώς αυτό να αποφύγουμε, να, ε, γεμίσουμε τις τρύπες δηλαδή, να καλύψουμε τα κενά. Τα BEPS μόνα τους μπορεί να φαίνεται ότι είναι έκφραση κοινή λογικής, αλλά στην πραγματικότητα δεν αρκούν. Είναι όμως δυνατό, κύριε Στασλή Φόξ, να σχολιάσετε για το λόγο, γιατί η πρότασή σας για τα υβριδικά είναι πιο χαλαρή από την πρόταση του ΩΣΑ. Σε κάποιε περιπτώσει, ναι, λέτε ότι είσαστε πιο αυστηρό, αλλά εδώ είστε πιο χαλαρό. Ναι, το, το έκανα, απαντάει ο κ. Μασουβισή. Για να λάβουμε υπόψη αυτά που αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αναγκαστήκαμε να προσαρμόσουμε τη δική μας ε, ε, πρόταση για να προσαρμοστεί με την ομολογία του δικαστηρίου. Τόσο απλό είναι. Και Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε όλα τα BEPS, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε και το BEPS, αν θέλουμε να είμαστε εξίσου αποτελεσματικοί όσο το BEPS σε διεθνέ επίπεδο. Και αυτό άλλωστε είναι καλό και για την διεθνή μας στρατηγική. Ευχαριστούμε τον κύριο Επίτροπο και τώρα εξ ονόματος της η κόρα Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μουσκοβισή που βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα και η δική μας ομάδα εκτιμά ιδιαίτερα το πακέτο που προτείνεται, το χαιρετίζουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε μαζί σας. Η διαφάνεια κατά πάσα πιθανότητα είναι το πιο σημαντικό μας όπλο. Όπως είπα όμως και στο Στρασβούργο, δεν φτάνει να κάνουμε ε, το σωστό, πρέπει να το κάνουμε και σωστά, ορθά να το εκτελούμε και ορθά. Γι' αυτό λοιπόν και έχω να σα θέσω κάποιε ερωτήσει. Το πακέτο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο έχει σήμερα, θα μπορούσε να προκαλέσει νομική αβεβαιότητα και διαφωνίε, γιατί κάποιε από του όρου δεν έχουν οριστεί με σαφήνεια. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη βάση της, ε, του κανόνα ΓΚΑΡ που προτείνεται για την καταπολέμηση των παραβιάσεων. Οι ε, διεθνεί εταιρείε σε ό,τι αφορά τις δράσεις τους ε, που έχουν ως σκόπο την προαποφυγή που δεν έχει να κάνει κάτι με την εμπορική πραγματικότητα θα μπορούσαν να θυμηθούν. Αλλά πώς ορίσετε το essential purpose, ε, valid economical reasons, ε, ο σκοπός, ο βασικός σκοπός ε, και η ορθή οικονομική λόγη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ορισμών σε ό,τι αφορά λοιπόν το παγκόσμιο προσκήνιο. Πέρα από αυτά που ρώτησε ο συνάδελφός μου από το ΕΛΚΑ, κατηγορήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπονομεύει την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα BEPS. Πείτε μας λοιπόν πώς απαντάτε συγκεκριμένα στην επιστολή αυτή και τελική ερώτηση. Η προτάσή σα δεν περιλαμβάνει μεταβατικέ ρυθμίσει προκειμένου οι επιχειρήσει να προσαρμοστούν εν αυτό το χρόνο. Θα το λάβει αυτό υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρχει αρκετό χρόνο και για τι επιχειρήσει και τα κράτη-μέλη για να προσαρμοστούν. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω σε, απαντώντας σε, ε, σε σχέση με την επιστολή από, την, το Υπουργείο Οικονομικών της ΕΠΑ εκτιμούμε ιδιαίτερα και η Κομισιόν θέτει το θέμα αυτό τη φοροαποφυγή στην κορυφή των προτεραιοτήτων. όλε οι επιχειρήσει ανεξάρτητα από το που προέρχονται, που έχουν και δημιουργούν κέρδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να καταβάλουν του εθνικά προβλεπόμενου φόρου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν μπορούν οι εθνικέ αρχέ να δίνουν φορολογικά προνόμια σε κάποιε μόνο επιχειρήσει που δεν τίθενται σε, όλη σε όλε τι επιχειρήσει. γιατί αυτό είναι ασύμβατο με το ευρωπαϊκό νόμο. Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν θα πρέπει να ζητήσει το, να ζητήσουν οι εθνικές αρχές από τις επιχειρήσεις τα ποσά τα οποία, από τα οποία απαλλάχθηκαν. Η απάντηση θα δοθεί από τον πρόεδρο Γιούγκερ αλλά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ισχύει για όλε τι επιχειρήσει που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση κατά των ε, Αμερικανικών επιχειρήσεων στην περίπτωση αυτή. Θα ενημερώσουμε λοιπόν τι ε, Αμερικανικέ Αρχέ για αυτό. Το έχουμε ήδη πράξει σε διάφορε περιστάσει. Θα δώσουμε τι απαραίτητε διευκρινήσει. Παρά το γεγονό ωστόσο ότι οι κρατικέ επιδοτήσει ε, δεν είναι στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Θα το συζητήσω αυτό με τον Τζακλού στη Σανγκάη την επόμενη εβδομάδα στο G20. Όσον αφορά, όσον αφορά τον ορισμό της ρήτας κατά των ε, καταχρήσεων για την καταπολέμηση της ε, πρόκειται για κανόνα ο οποίος λειτουργεί ως δίκτυα ασφαλείας. Δηλαδή όπου δεν προβλέπονται ρητά κανόνες, ε, κοιτάει τη σκοπιά της αφέμητης φοροαποφυγής. Και άρα έχουμε ένα στοιχείο ουσιώδες εδώ των μέτρων, των συγκεκριμένων μέτρων κατά των καταχρήσεων. Αυτό το γενικό μέτρο θα κοιτάει να αντιμετωπίζει καταστάσεις για τις οποίες έχουμε αδυναμία δράσεως προς το παρόν. Είπατε και εσείς ίδια, είναι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις για το δικαστήριο επανειλημμένως έχει εκφραστεί μέσω της νομολογίας του και έχει δώσει συγκεκριμένους ορισμούς και διατάξεις, πράγμα το οποίο έχουμε και μέσα στην οδηγία Murphy. Και εν τέλει για το χρονοδιάγραμμα, όπως και με τον ΩΣΑ, Όλα τα μέλη του ΩΣΑ μάλιστα θα πρέπει να το τηρήσουν. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει την κατάρτιση της νομοθεσίας τους με βάση αυτές τις προτάσεις μας και ως εκ τούτου ακολουθούμε την βάση των συμφωνιών BEPS και κλείνοντας ευχαριστώ πολύ την ομάδα σας για την υποστήριξη που εν γέννη εκφράζει προς τη δική μας προσέγγιση. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις αντιδράσεις των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστημά μας στο δίκαιο του ανταγωνισμού και των κυρώσεων, γιατί δεν έχουν κάτι αντίστοιχο στην νομοθεσία τους για τις κρατικές ενισχύσεις. Και η Federal Trade Commission, η αντίστοιχη επιτροπή για το θεμητό ανταγωνισμό, και το εμπόριο δεν έχει λειτουργίε και αρμοδιότητε αντίστοιχε με τι Ευρωπαϊκέ Επιτροπέ στον Ανταγωνισμό. Εμεί θα επισκεφθούμε τι ΗΠΑ το Μάρτιο για να συναντήσουμε ε, ομολόγους μας από τις ε, Επιτροπές Αρμόδιες για τα Οικονομικά και τα Φορολογικά, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το, ε, τη Γερουσία και θα κοιτάξουμε να κάνουμε επαφές, να τους προτείνουμε επαφές ε, σε σχέση με τις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Γιατί είδαμε με έκπληξη πέρυσι ότι η τα διευθυντικά θελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων όταν πήγαιναν στο Καπιτόλιο για να δώσουν μαρτυρία ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων είχαν διαφορετική στάση από αυτήν την οποία ακολουθούσαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον εμείς τους καλούσαμε και γι' αυτό ίσως θα ήταν σκόπιμο να οργανώσουμε κοινέ ακροάσει με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πραγματικά ποια είναι η θέση αυτών των επιχειρήσεων. Εκ μέρου τη ΓΚΟΕ, ο κύριο Μπιέγκα. Είχα μία σειρά ερωτήσεων, συγκεκριμένων ερωτήσεων. Σε σχέση με την έκθεση, την αναχώρα έκθεση προβλέπονται 750 δις ευρώ. Αυτός είναι ο κύκλος εργασιών, αυτό είναι το κατόφλι για τον κύκλο εργασιών που αφήνει μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων εκτός. Δεν θα ε, μπορούσαμε να έχουμε ένα κατώτερο κατόφλι έτσι ώστε να μην ε, αποφεύγουν αυτή τη βάση οι επιχειρήσεις. Σε σχέση με την μελέτη αντικτύπου που θα γνωρίσουμε τον Απρίλιο, θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο θα διενεργηθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ή έχει ανατεθεί σε μια εξωτερική ε, εταιρεία μελετών. Και αν ναι, ποια είναι αυτή. Θα είναι η PwC που διενέργησε μια παρόμοια μελέτη στην περίπτωση του τραπεζικού συστήματος. Σε σχέση με τη φορολογική βάση τώρα, η ΟΣΑ προβλέπει ε, ένα χάσμα, μία διαφορά 10 με 30%. Εσείς αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε ένα ανώτερο όριο, δηλαδή μια υψηλότερη ποσόστια αναλογία. Πώς ε, ορίζεται λοιπόν αυτό το πλαίσιο για την αφαίρεση των τόκων. Και σε αυτή την περίπτωση γιατί αποκλείσατε τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις από αυτή την ε, διάταξη. Σε σχέση τώρα με τις ε, επιχειρήσεις, τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις που βρουν στο εξωτερικό θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο κριτήριο φορολόγησης αυτών των επιχειρήσεων, δηλαδή σε μία τρίτη χώρα η ποσοστή αναλογία φορολόγησης που θα ισχύει για το εξωτερικό θα είναι της τάξης του 40%. Ισχύει γιατί αν σε μια χώρα υπάρχει ένα 30% θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η φορολογική βάση σε μια συγκεκριμένη χώρα ε, αντικατοπτρίζει αυτή την ποσοστή αναλογία γιατί υπάρχουν διαφορετικές φορολογικές βάσεις 20, 30, 40% γιατί εσείς επιλέξατε μία ε, ποσοστία αναλογία και επίσης δεν θα έπρεπε μέσα στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο να ισχύουν αυτά τα μέτρα τη στιγμή που οι φορολογικοί παράδεισοι υπάρχουν εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Θα ήθελα να πω, το είπα άλλωστε αμέσως στον κύριο Φόξ, ότι μένουμε στη βάση των BEPS του όσα προδιαγραφές σύμφωνες με αυτές του ΩΣΑ, 750 εκατομμύρια ευρώ που ορίζει και όσα, με στόχευση τις πολυεθνικές εταιρείες εκείνες οι οποίες έχουν τα μέσα να προχωρήσουν σε επιθετικό φορολογικό προγραμματισμό και μέτρα ή μηχανισμούς βελτιστοποίησης της φορολογίας τους. Εμείς μπορούμε να παρακολουθούμε, να προσκολόμαστε ούτως υπήν ως Επιτροπή στον ΩΣΑ, αλλά προχωρούμε και λίγο περισσότερο. Για, τα, για τις μελέτες τώρα. για τη δημοσιοποίηση του ΣΥΜΠΙΣΙΑ που είναι δουλειά του συναδέλφου Τζόναθαν Χίλα των δικών του υπηρεσιών. Θέλω να σας επισημάνω ότι αυτές οι μελέτες είναι κυρίως εσωτερικού χαρακτήρα. Οι κανόνες CFC εφαρμόζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής και για την ε, ε, αφαίρεση των ε, κερδών έχουμε το ανώτερο ίσως ποσοστό, αλλά ε, μπορούν τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν ακόμη πιο απαιτητικού κανόνε Οι χρηματοπιστωτικέ εταιρείε προ το παρόν αποκλείονται, συνεχίζονται όμω αντίστοιχα οι εργασίε του ΩΣΑ και μπορούν να οδηγήσουν νέε εξελίξει. Όπω είπαμε, αυτό ο αγώνα δεν σταματάει για την καταπολέμηση της φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, επιθετικού φορολογικού προγραμματισμού, Όπω δεν σταματάει στην Επιτροπή, δεν σταματάει και στον ΩΣΑ. Είμαστε σε ένα στάδιο μόνο αυτή τη πορεία. αλλά θα συνεχίσουμε. Οι πράσινοι Κυρία Ευαζολή, Πρόεδρε ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο οικολόγοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δημοσίευσαν μια έκθεση για τις πρακτικές βελτιστοποίησης φορολογίας της επιχείρησης IKEA. Παρά περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στα οικονομικά του ομίλου έχουμε μπορέσει να αξιοποιήσουμε, να υπολογίσουμε σε ένα δις ευρώ επί έξα ετία το διαφυγόν έσοδο για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Πολλά ήταν τα ρήγματα και τα κενά στη φορολογία που ενθάρρυναν τα κράτη-μέλη τα ίδια, οι κάτω χώρες, το Λουξεμβούργο σε ένα βαθμό, επιτρέπουν έτσι την μη φορολόγηση του ε, τόκου επί των μερισμάτων και των royalties, των πνευματικών δικαιωμάτων των ε, χρήση. Και έτσι, και σε ένα βαθμό βέβαια και το Λίχτενστάιν, και έτσι βρέθηκε σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση το Λουξεμβούργο σε σχέση με την έκφραση ορισμένων ενιών και αντιλήψεων σε σχέση με τη φορολογία. Βεβαίω, το πακέτο που προτείνεται αποτελεί ένα σημαντικό ε, στάδιο, αλλά δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αποδιαρθρώσει κάποιες φορολογικές πρακτικές όπως αυτές που ακολουθεί η επιχείρηση IKEA και άλλες. Χρειάζεται μια ελάχιστη φορολόγηση, κοινή φορολόγηση ή μια εναρμόνιση της φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε ε, Επίτροπε, μπορείτε να επιβεβαιώσετε πρώτον ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των τελών Ιανουαρίου ε, δεν θα επέτρεπαν το όντι να τεθεί ένα τέρμα στο σύστημα IKEA όπως το ονομάζουμε και το χρειάζονται εκ τούτου και άλλα μέτρα. Δεύτερον, ότι η ε, έννοια, η διαφοροποίηση ως προς την έννοια την φορολογική στο Βέλγιο οδηγεί σε σημαντικές ε, απώλειες εσόδων και ως εκ τούτου πρέπει να εξεταστεί με τρόπο άτεγκτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι ε, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν οι συμφωνίες έτσι ώστε να προχωρήσουμε το έχετε δυνατό σε επίπεδο συμβουλίου σε ενιαίο, ελάχιστο έστω, κοινό φόρο. Τι θα κάνετε για να προσφατεύσετε και να υπερασπιστείτε τα κράτη-μέλη. Ο Κυρία Ζολή, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και τους πρασίνους για αυτή την έκθεση και φυσικά ε, ε, χαίρομαι που βρίσκεται θετικά σημεία και στη δική μας προσέγγιση. Μετά από την ε, ε, δημοσίευση αυτή της έκθεση μας ενδιαφέρει το θέμα της απαλλαγής στη βάση όπως ισχύει στο ε, προτιμησιακό καθεστώς για τις αμοιβέ και του patent box και ε, την περίπτωση του Λίχτενστάιν, ας πούμε μιας χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν υπάρχουν αυτά τα μέτρα για τη βελτιστοποίηση της φορολογικής αντιμετώπισης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτή την οδηγία για να αλλάξει η φορολόγηση στη χώρα προέλευσης, τη στιγμή που δεν γίνεται σωστή φορολόγηση. Υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση. Τα κράτη-μέλη θα ε, αλλάξουν το pattern box όπως ορίζεται από τον Όσα και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της ε, σωστής φορολογικής συμπεριφοράς. Παρακολουθούμε την εξέλιξη. Όσον αφορά τις ε, σχέσεις με τις τρίτες χώρες, το πακέτο της 27ης Ιανουαρίου ορίζει τις ελεγχόμενες εταιρείες αλλοδαπής προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια της ε, χρηστής ενισχυμένης διακυβέρνησης και έχουμε ένα πρότυπο ανταλλαγής ε, πληροφοριών σε σχέση με τους ε, πραγματικούς ε, δικαιούχους. Στην περίπτωση του Λίχτενστάιν υπογράψαμε μία διμερή συμφωνία για την άρση του τραπεζικού απορρίτου και τώρα γίνεται μία συζήτηση για τα φορολογικά καθεστώτα που ισχύουν. Όπως ξέρετε και με το Σαν Μαρίνο και με την Ανδόρα και στο Σαν Μαρίνο θα βρεθώ για να υπογράψουμε μια παράλληλη διμερή συμφωνία. Το πακέτο της 27ης Ιανουαρίου με βάση ε, και παράλληλες πρωτοβουλίες αποτελεί επαρκή απάντηση σε σχέση με την έκθεση και εάν όμως μετά από λεπτομερή μελέτη φανεί ότι δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των ε, φαινομένων, εγώ φέρω την ευθύνη να βελτιώσω τα κατάλληλα μέσα για να μην υπάρχει ε, διαφοροποιημένη φορολογική βάση η οποία να πλήττει ορισμένα κράτη. Μιλήσατε και για την περίπτωση των ρητρών ε, κατά της κατάχρησης και στην περίπτωση του Βελγίου θα πρέπει να γίνει ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να καταχρώνται αυτό το σύστημα. Και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση και σας ευχαριστούμε για αυτήν την έκθεση που ήταν άκρος χρήσιμη. Και εγώ συμμερίζομαι ε, τις ευχαριστίες ε, του ε, Επιτρόπου και όπως ξέρετε προβλέπουμε ακροάσεις σε σχέση με μικρά κράτη και Έχουμε καλέσει στο Λίχτενστάιν τις επόμενες εβδομάδες για να το αντιμετωπίσουμε. Ο Μάρκο Βάλι έχει το λόγο από την Ευρώπη της Ελευθερίας. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ερωτήσεις προς τον Επίτροπο. Καταρχήν, ως προς τις μακροοικονομικές ε, ανισότητες. Ξέρετε ότι η Ολλανδία χρησιμοποιεί τις σταθερές ε, ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες για να προβεί σε κέρδη και φυσικά και τα tax rulings και τις φορολογικές συμφωνίες αυτού του τύπου. Νομίζω λοιπόν ότι οι συστάσεις θα πρέπει να προβούν σε κυρώσεις κατά αυτών των χωρών και όχι να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δέχεστε αυτή την θεώρηση των πραγμάτων ή δεχόσαστε αυτό το παράδοξο, δηλαδή ε, μιλάμε για μια επιτροπή Juncker που εκπροσωπεί το Λουξεμβούργο όπου ε, υπήρξε πληθώρα tax rulings με φοροαποφυγή και από την άλλη πλευρά πλεονάσματα στον φορολογικό ισολογισμό σε σχέση με τα κέρδη και τις πηγές των κερδών. Είπατε ότι αυτή η πόρτα είναι κλειστή θα πρέπει να ξέρετε ποιος κλείνει όμως αυτές τις ε, πόρτες. Μπορούμε να έχουμε ονόματα για να ξέρουμε ποια είναι τα κράτη που φέρουν ευθύνη. Έτσι ε, ε, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις χώρες που παραβιάζουν αυτό το πλαίσιο. Επίσης πολλά αναφέρθηκαν στον τύπο για την διαφάνεια και για, τον κανόνα, για τους κανόνες συμπεριφοράς. Σε αυτά τα έγγραφα υπάρχουν πολλά σκοτεινά τμήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στα πάντα ή ορισμένοι αντιτάσσονται σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν υπάρχει πλήρης πρόσβαση στα, έγγραφα αυτά, δεν είναι πλήρως ε, δημόσια. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ε, δεν θα ήθελα τώρα να σχολιάσω τις εκθέσεις αναχώρα, γιατί όπως ξέρετε η Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα θα, διαβουλευθεί, θα προβεί σε διαβουλεύσει από το θέμα τους και δεν θα ήθελα τώρα να επεκταθώ για τις εκθέσεις αυτές. Μιλήσατε για τις μακροοικονομικές ανισότητες που γνωρίζουν ορισμένες χώρες. Η Ευρωζώνη έχει ένα τρέχον πλεόνασμα, είναι γεγονός το οποίο είναι μεγάλο. Και έχουμε να κάνουμε με χώρες που πρέπει να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες, αλλά η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν υψηλά πλεονάσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα περιθώρια ελιγμών τους για επενδυτικά σχέδια. Αυτό θα υπενθυμίσουμε και φέτος. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ε, αυτά που ε, αναφέρατε κατά του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας. Η Λουξεμβουριανή ε, Προεδρία ήταν εξαιρετική και όπως ξέρετε εγκρίναμε και την οδηγία για τις φορολογικές συμφωνίες τύπου tax ruling υπό Λουξεμβουριανή Προεδρία και η Ολλανδική Προεδρία ε, είχε μια, έκανε μια καλή αρχή και πιστεύω ότι ο Γερούν Ντάισεμπλουμ θα προχωρήσει πολύ γρήγορα και πολύ μακριά. Αυτή η συζήτηση είναι μια δημόσια συζήτηση. Προσπαθούμε να ορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές και με βάση τα BEPS και όπως είπε η Ολλανδική Προεδρία θα έχουμε ένα συνολικό έγγραφο για να δούμε τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια και τι διαφοροποιήσεις θα γίνουν σε σχέση με μια πρόταση για τη φορολογική βάση. Όλα τα κράτη-μέλη συνεργάζονται για να φορολογούνται τα πραγματικά κέρδη εκεί που ε, γίνονται, εκεί που προκύπτουν, σε σχέση με την δημοσιοποίηση τώρα των εγγράφων, ορισμένα έγγραφα δεν μπορούν να είναι ε, δημόσια. Εμείς ε, δεν φέρουμε ευθύνη γι' αυτό, θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια μέχρι τέλους. Αλλά επαναλαμβάνω, οπωσδήποτε τα πρακτικά θα είναι στη διάθεσή σας στην κάμερα βέβαια έτσι ώστε να γνωρίσετε ορισμένα στοιχεία τα οποία σήμερα, μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, Επιτροπέ Κομοσκοβησή. Στις 28 Ιανουαρίου μας παρουσιάσατε το πακέτο το σχετικό το οποίο συζητάτε σήμερα και πραγματικά βασίζεται σε τρεις πυλώνες της ε, εγγυώσης ε, σύμφωνα με τις ε, υφιστόμενες ε, ρυθμίσεις σε πιο δίκαιη ε, συνθήκες ανταγωνισμού και μεγαλύτερη διαφάνεια μαζί με μια εξωτερική στρατηγική σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση πολυεθνικών ομίλων. Βάση του πακέτου αυτού είναι η πρωτοβουλία BEPS του ΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης ε, και μεταφοράς των κερδών. Και είπατε σήμερα, κυρία Επίτροπε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να είναι κινητήριος δύναμη για την εφαρμογή των ε, BEPS αυτών. Θα ήθελα να συζητήσω και την επιστολή αυτή, η οποία αναφέρθηκε ήδη σήμερα του Υπουργού Οικονομικού, Οικονομικών των ΗΠΑ προς τον ε, κύριο Γιούγκερ. Με εσάς σας ενημένω, κυρία Επίτροπε αληθεύει αυτή η κατηγορία που περιέχει σε ό,τι αφορά δηλαδή τα μέτρα εφαρμογής που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συνάδουν με τις πρωτοβουλίες ΠΕΠΣ e Με την πρωτοβουλία αυτή με την οποία διατείνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέλει να προωθήσει ως κινητήριος δύναμη και που ε, δεσμεύει τα 27 κράτη-μέλη για συντονισμένη εφαρμόγη και η Γερουσία στην Αμερική ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, στη Σχετική Επιτροπή συζητήθηκε το θέμα αυτό και ο Υπουργό Οικονομικών συστήνει στην Επιτροπή να ανασταλούν οι σχετικές ε, έρευνες από την Επιτροπή Φριστάγκεν. Ερωτώ λοιπόν, πώς το δικαιολογείτε αυτό. Πώ δικαιολογείται το γεγονό ότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στην πράξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των μέτρων δηλαδή αυτών που συστήνονται στα ΠΕΠΣ e και στις δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν συνάδει με αυτά. Που υποτίθεται ότι αυτά ακριβώ τα ΠΕΠΣ e αποτελούν τη βάση για το προλογικό πακέτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Επίτροπος να απαντήσει τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάπλη. Θα περιοριστώ στην υπενθύμηση αυτού που είπε και ο Πρόεδρος και ο υποφαινόμενος σε προηγούμενη απάντηση ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντικές σε οικονομικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως και σε επίπεδο φορολογικής συνεργασίας επίσης. Το είπα και νωρίτερα. Εάν δεν είχαν και υποστηρίξει και οι ΗΠΑ για να μην πω ότι είχαν την πρωτοβουλία των συμφωνίων BEPS, δεν θα είχαν καν προχωρήσει, ίσως να μην υπήρχαν καν οι συμφωνίες για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή των πληροφοριών. Ο Τζακ Λου, ο Υπουργό των Οικονομικών, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και βεβαίω υπάρχει η επιστολή που απευθύνθηκε στον πρόεδρο Γιουνκέρ και όχι σε κάποιο επίτροπο και θα λάβει την απάντησή της. Αλλά είπε ο κύριος Λαμασουρίδη ότι τα δικαιοδοτικά μας συστήματα δεν είναι ταυτόσημα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα αυτά έναντι των επιχειρήσεων δεν είναι ο ίδιος. Υπάρχουν όμως ε, φορείς ιδιωτικού δικαίου που έχουν όχι συστημικά πάντως λάβει κάποιες, ε, κάποια μέτρα, κάποιες διατάξεις που έπληξαν πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση βάρος των πολυεθνικών, των Αμερικανικών. Θα πρέπει να συνεχιστεί και η φορολογική όπως και η οικονομική συνεργασία. Αυτή λοιπόν η απάντηση θα δοθεί. Θα συνεχίσουμε το διάλογο με τις αρχές των ΗΠΑ και σας είπα και εγώ θα είμαι στη Σανγκάη τις μερικές μέρες στο G20, θα δω το Τζακλου και θα συζητήσω μαζί του πώς μπορούμε να συνεχίσουμε προς μια καλή συνεργασία είπαμε ότι στην υπόθεση αυτή, όπως πάντα, είμαστε αλληλέγγυοι με τη συναδελφό Βεστάγκερ από την ε, Γενική Διεύθυνση του Ανταγωνισμού, όπως και εκείνη στέκεται στο πλευρό μου στα θέματα τα φορολογικά. Είμαστε μια διανδρία θα έλεγα. Εγώ προτείνω νομοθεσία, εκείνη την εφαρμόζει με τρόπο στεναρό. Ξέρετε είναι μια πολύ θαραλέα γυναίκα. Κάνει τη δουλειά της με πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα, θα το ξαναπώ, πολύ καλή πολιτική προσέγγιση η οποία δεν εμπνέεται από καμία μορφή διακριτική μεταχείριση. Ευχαριστώ, κύριο Χοκμάρκ, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσά, κύριε Επίτροπε. Καταρχά, θα ήθελα να πω ότι αντέδρασα κάπω όταν αναμίξατε την φοροαποφυγή με τι μολυθνικέ εταιρείε και κατά πόσο να ακολουθούν ή δεν ακολουθούν τον νόμο. Τα θέματα αυτά θα τα θα τα κρίνει το δικαστήριο, όχι δεν θα κρυφθούν από πολιτικές δηλώσεις. Κατά δεύτερον, πολλά ερωτήματα ε, τέθησαν για τη μελέτη αντικτύπου, για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά. Η διαφορά δεν είναι το τι θα πρέπει να κάνουμε, πιστεύω. Το θέμα είναι το πώς θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και έχουμε λοιπόν τις συστάσεις του ΩΣΑ είναι σαφέστατο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θέλει να υπερβεί ακόμα και τις συστάσεις αυτές και αυτό ασφαλώς έχει και συνέπειες. Μου κάνει λοιπόν κάπως εντύπωση το γεγονός ότι δεν άκουσα εδώ στη συζήτηση αυτή τις λέξεις ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις, έλλειμμα επενδύσεων μάλλον και που θα πρέπει να καλυφθεί. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Αυτό είναι το σημαντικό, το αποφασιστικό στοιχείο Ένα από τα προβλήματα λοιπόν που έχει η Ευρώπη ότι έχουμε πιο υψηλό γενικό φόρο από ότι οι υπόλοιπε περιοχές του κόσμου. Αν λοιπόν ε, δράσουμε με τον λάθος τρόπο θα υποφέρουμε ακόμα πιο πολύ. Θα καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και τις απάτες ε, της φορολογικές και τις ε, επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν τους πόρους τους. Αυτό δεν μπορούμε να το αποταχθούμε, αλλά είναι σημαντικό να δείξει συνέπεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πολιτικές ανάπτυξης για να καλυφθεί το χάσμα των επενδύσεων και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και το να ξεπεράσουμε τις ε, συστάσεις του ΩΣΑ αποτελεί ένα ρίσκο μήπως θα καταλήξουμε να έχουμε υψηλά, υπερβολικά υψηλό φορολογικό φορτίο, ακόμα πιο υψηλό από τη σήμερα σε σύγκριση με τη ΣΥΠΑ. Αυτό θα υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα. Εγώ αυτά τα θέματα θέλω να αντιμετωπίσετε, γιατί θα είναι ζωτική σημασία για την καταπολεμήση της φοροαπάτης και της φοροαποφυγής. Σας ευχαριστώ, ο Επιτροπός. άλλο πράγμα η φοροαπάτη και άλλο πράγμα ο φορολογικός σχεδιασμός. Αλλά όταν οι επιχειρήσεις ενεργούν γνωρίζοντας ακριβώς που βρίσκονται τα παραθυράκια και τα εκμεταλλεύονται, έμα στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, διότι το αποτέλεσμα είναι απώλειες για τους δημόσιους προπολογισμού λιγότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων αυτών και πολύ μεγαλύτερη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε που έγινε οι διαφορές και στο πακέτο μας ακριβώς αυτό θέλουμε και εμείς να καταπολεμήσουμε. Την ε, φοροαποφυγή, την φοροαπάτη, την ε, διάβρωση της φορολογικής βάσης και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε με αυτά και συμφωνώ με αυτά που αναφέρατε. Για την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα δε, αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο επέμεινα επανελειμμένα στα εισαγωγικά μου σχόλια και σκοπεύω να το πράξω εκ νέου. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι σύμφωνα με την προσέγγιση εφαρμογή των συστάσεων αυτών θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα έχουμε και λιγότερη γραφειοκρατία και πιο πολύ νομική βεβαιότητα, μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα για τις ε, επιχειρήσεις μας στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές ε, ε, διαφορετικές επικράτειες που έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή των ε, BEPS του ΩΣΑ. Είμαστε δεσμευμένοι να καταπολεμήσουμε λοιπόν ε, την φοροαποφυγή. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Πάντα θέλουμε να συνδυάζουμε τις δύο αυτούς τομείς διαφάνεια μένα από τη μία και καταπολέμηση ε, της φοροαπάτης και της ε, διαφυγής στον φορολογικό σχεδιασμό. Το πώς το πράττουμε αυτό έχει συζητηθεί από μακρόν στους κόλπους του ΩΣΑ. Δεν προτείνουμε κάτι καινούριο, κάτι άγνωστο στα κρατημέλη, όλα αυτά έχουν συζητηθεί. Και το θέμα της ανταγωνιστικότητας και των ίσων όρων ανταγωνιστικότητας μεταξύ των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων ε, χωρών. Και οι μελέτες καταδεικνύουν ότι 30% παραπάνω πληρώνουν οι μικρές επιχειρήσεις σε φόρο. Και Νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές Δημοκράτες, ο κύριος Κόφουρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Επιτροπέ, καταρχάς θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για το φορολογικό πακέτο και για την σαφή σας τοποθέτηση για τις εκθέσεις αναχώρα. βλέπουμε στη συνέχιση της συζήτησης αυτής. Ένα αρχικό σχόλιο και προς τον ε, καλό συνάδελφο Γκούναρ Χορκμάρκ. Πιστεύω ότι είναι γεγονός ότι η φόρα αποφυγή των μεγάλων ε, ομίλων απειλούν, ε, απειλεί και τον ανταγωνισμό και το κράτος πρόνοιας και το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες φορολογούνται 30% παραπάνω από τις πολυεθνικές είναι ανησυχητικό. Το θέμα λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά να διασφαλίσουμε την δικαιοσύνη και τον ισονταγωνισμό. Αλλά να πω και ένα ακόμα πράγμα και να σας θέσω και μία ερώτηση. Πολλές παλαιστινικές εταιρείε από ό,τι ξέρετε έχουν ως σκοπό τη μηδενικό προλογικό συντελεστή και βοηθούνται από μεγάλες συμβουλευτικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά εντρήματα. Και έτσι φτιάχνουν περίπλοκα και αμφιλεγόμενα ε, ύποπτα ε, φορολογικά καθεστώτα, φορολογικούς παραδείσους. Και αυτό το αντιμετωπίσαμε λοιπόν στην Επιτροπή Τάξη. Και θέλουμε να υπάρξει δράση κατά των τακτικών αυτών. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να δοθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα προβλέπει υπαρκείς κυρώσεις κατά των επιχειρήσεων, των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών εντρημάτων, των υπηρεσιών, των εταιριών συμβουλευτική, όλου αυτού του συναφιού που εμπλέκεται στις πρακτικές φόρο διαφυγής. Νομίζω ότι είναι ύψης της σημασίας να υπάρχουν κυρώσεις κατά αυτόν. Γιατί αν προωθεί κανείς τέτοιες πρακτικές ε, ε, επιθετικής φορολογικής ρύθμισης, ε, πιστεύω ότι χρειάζονται κυρώσεις. Και νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ακόμα και ε, άρσης της ε, άδειας λειτουργίας τους. Υπάρχει λοιπόν οποιαδήποτε πρωτοβουλία προ την κατεύθυνση αυτή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να χτυπήσουμε το κακό ρίζα του. Ευχαριστώ κύριος Επίτροπο. Έχει το λόγο για να απαντήσει. ο αγώνας κατά των καταθέσεων στα φορολογικά ξεπερνάει αυτά τα οποία έχουμε μαθεί τώρα προτείνει. Πρέπει να είμαστε ωστόσο ε, σαφείς και να έχουμε συνέντευξη όμως ότι είναι περίπλοκο και κοινωνικά το θέμα της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και ίσως μπορεί να ξεπερνάει κάθε μηχανισμό προγραμματισμού και οργάνωσης φορολογικής. Ξεκινούμε όμως αυτή την προσπάθεια με την δέσμη μέτρων που σας παρουσιάζω. Θα συνεχίσουμε, είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό. Θα δούμε πού και πώς θα προχωρήσει το θέμα του country reporting, των εκθέσεων ανά χώρα. Είμαστε αισιόδοξοι, σας το είπα, αλλά δεν θα σταματήσουμε σε αυτό. Υπάρχει μια πολιτιστική, ψυχολογική, πολιτική μετάλλαξη που εξελίσσεται και δεν πρόκειται να σταματήσει και θα την παρακολουθήσουμε. Και αυτό σημαίνει ότι, μπορούμε να, ότι ενδέχεται να προχωρήσουμε περισσότερο ακόμη στον τομέα που σας ενδιαφέρεται. Που σας ενδιαφέρει. Για τους ε, λογιστικούς ελέγχους, Φερρυπίν, της προτάσεις του 2014, θα εξετάσουμε τις ε, συνέπειές τους και την αποδοτικότητά τους σχέση με τις επιχειρήσεις πριν καταθέσουμε νέες προτάσεις. Ο κύριος Δάριος Ρωσάτη. Μόνο μια συμπληρωματική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Μια πολύ σύντομη ερώτηση, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Γιατί είδαμε με τα τάξη rules προκατακτικές ε, φορολογικές συμφωνίες και την ε, ανάληψη δράση από την Επίτροπο Φέρσταγκερ κατά των κατοχωρών του Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Θεώρησε ότι ήταν παράνομες. Όταν δημοσιεύτηκαν αυτές οι συμφωνίες, ε, οι δράστες αυτής της παρανομίας, χώρες δηλαδή αφενός επιχειρήσεις αφετέρου, ευνοήθηκαν και μάλιστα οι χώρες από το αυξημένο φορολογικό έσοδο. Ε, ρωτώ λοιπόν κύριε Μοσκοβισή, ποια είναι η ευθύνη του κάθε επιτρόπου εν προκειμένου. Όταν μια χώρα ε, προβαίνει σε μια τέτοια φορολογική συμφωνία θα πρέπει να μην επιβραβεύεται, αλλά να τιμωρείται. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το αντιμετωπίσετε αυτό. Πώς θα το χειριστείτε. Σας ευχαριστώ. Ένα πιο διαφανές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις πιστεύω θα διευκολύνει αυτή τη μετάβαση. Είναι ένα ζήτημα άλλωστε και ιδιών πόρων που μπορούμε να συζητήσουμε. Ξέρετε ότι με τον Αλένα Μασούχ είμαστε στην ομάδα για τους ιδίους πόρους. Εκπροσωπείται και κύριος, ε, εκπροσωπείται όλη η Επιτροπή, γιατί είναι και ο κύριος Γιουνκέρ και ο κύριος Τούμερμανς και τα λοιπά. Και η κυρία Βεστάγκερ μέσα σε αυτήν την ομάδα. Ο κύριος Λαμασούρ, ναι, θα είναι κομμάτι των συστάσεων, αγαπητέ φίλε, Κόφαουτ. Και στην ε, σύσταση της τάξε το έχουμε ήδη αναφέρει. Θα επανέλθουμε λοιπόν Λογικό είναι σε τελευταία ανάλυση. Και δεν θα είναι, δεν θα είναι πρόστιμο, αλλά υπενθύμηση φόρου. Υποχρέωση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλλει ε, την, ε, το μέτρο αυτό έτσι ώστε να εξισορροπήσει την απώλεια εσόδων την οφειλόμενη στον, στη στρέβλωση του ανταγωνισμού του φορολογικού. Ο κύριος Ρωσάτη που τώρα βλέπουμε ότι είναι ελεύθερος να μιλήσει. Παρακαλώ. Επιτροπέ, να επανέλθω στο θέμα το, της δημόσιας πρόσβασης στις εκθέσεις αναχώρα. Σας ρωτώ, ποια είναι η απόψή σας για τον αντίκτυπο, αν περάσει αυτή η λύση, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος σε ό,τι αφορά την συγκριτική θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ΕΠΑ, στην Κίνα. Η λύση αυτή για την αποκάλυψη των φορολογικών αυτών στοιχείων θα βάλει σε μειονεκτική θέση τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με τις 45 επιχειρήσεις. Και η άλλη ερώτηση που ανακύπτει. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία αυτή. Γιατί στην παρούσα φάση, αν σωστά καταλαβαίνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για το διαδικαστικό κομμάτι. Θα ήταν σωστό και προτιμητέο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει και δικαίωμα πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Θα βοηθούσε, θα είναι ωφέλιμο αν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δρούσε η Επιτροπή και ως θεματοφύλακα στις ε, οδηγίες. Σε ό,τι αφορά τώρα πάλι το θέμα της μέρης αντικτύπους, ο απότερος στόχος εξ όσων καταλαβαίνω του όλου εγχειρήματο είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πολυεθνικές θα πληρώνουν το ποσοστό που τους αναλογεί σε φορολογία στην Ευρώπη. Αυτό, αν τα καταλαβαίνω, σημαίνει ότι σε τελική ανάλυση θα πρέπει να πληρώνουν πιο πολλούς φόρους. Υπάρχει οποιαδήποτε εκτίμηση, αξιολόγηση του αντικτύπου που θα είχε αυτό στις επιχειρήσεις αυτές, στις εταιρείε αυτές. Υπάρχει κίνδυνος να σηκωθούν και να φύγουν κάποιες από αυτές τις εταιρείε και να πάνε σε άλλες επικράτειες λόγω των βελτιώσεων του συστήματος φόρου στην Ευρώπη. Καταρχάς, να επαναλάβω ότι αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ότι παρουσιάζουμε το πακέτο για την αποφυγή φοροδιαφυγής. Και είναι μια διαδικασία αυτή σε δύο βήματα. Σε πρώτη φάση και όπως είπατε, εφαρμόζουμε απλά τα πρότυπα, τα οποία ήδη έχει προτείνει όσα και θα περιοριστούμε στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και αρχών. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μοναδικό σωστό και θα πρέπει να γίνει. Αργότερα, τον Απρίλιο από τον Απρίλιο και μετά, θα πρέπει να καταθέσουμε και μία πρόταση για την δημοσίευση του CBCR. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί αυτή η πρόταση. Αυτό, όπως σας είπα, εξαρτάται από τα απορίσματα της μελέτης αντικτύπου, τα οποία δεν μου είναι γνωστά ακόμα, την οποία και διαξάγουν οι συνάδελφοι, οι υπηρεσίε του συναδέλφου. Όπως σας είπα, θα ακολουθήσουμε μια ρεαλιστική ε, προσέγγιση. Ακριβώς είναι το θέμα το οποίο θίξατε. Εγώ είμαι υπέρ. Α, και άλλοι υπέρ, αλλά θα δούμε. Για να μην διαμορφωθεί όμως ένα εχθρικό κλίμα προς τις εταιρείε. Και η απάντησή μου θα είναι αρκετά ξεκάθαρη. αν ο αντίκτυπο, ο οποίο φυσικά είναι δύσκολο να υπολογιστεί, θα είναι σημαντικό δεν θα πρέπει να ε, γίνει το βήμα αυτό τώρα. Αν φανεί ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα μεταξύ διαγνωστικότητα και διαφάνεια, θα μιλήσουμε γρήγορα. Πιστεύω ότι η ίση όρη λειτουργίας συνάδουν με τη δουλειά που γίνεται για την καταπολέμηση της διπλής φορολόγησης και αυτό θα μπορούσε να αντισταθμίσει την απώλεια ανταγωνιστικότητας. Σε ό,τι αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαι πάντα υπέρ μεγαλύτερου ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τέτοια θέματα. Αυτό κερδίσαμε και από την οδηγία για το tax rulings. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να συμμετάσχει σε συζήτηση μεταξύ δύο κρατών μελών. Αλλά το θέμα του κατά πόσο θα πρέπει να αποτελεί θεματοφύλακα της οδηγίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλό θέμα. Είναι καλό ερώτημα. Και σίγουρα θα χαιρέτιζα κάποια υποστήριξη από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ την κατεύθυνση αυτή. Αυτό θα ήταν καλό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κυρίω για το κοινό συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, ο Μορέλα, από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι, όπως είπαν όλοι οι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα. Φυσικά γίνεται πρόοδο και ε, έχει συμμετάσχει άμεσα σε αυτή τη διαδικασία και ο Επίτροπος Μοσκοβισή. Μιλάμε για ένα πιλιοτικό άλμα για την καταπολέμηση της φοραποφυγής. Νομίζω ότι είσαστε υπεραισιόδοξος ως προς τη θέση του Συμβουλίου. Ε, μιλήσατε για τη Λουξεμβουριανή Προεδρία που ήταν πολύ φιλόδοξη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Λουξεμβούργο έκανε μία φιλόδοξη πρόταση το Δεκέμβριο πριν να αποχωρήσει από την Προεδρία και τον Ιανουάριο δεν προχώρησε αυτή η, πρόταση γιατί είναι της αρμοδιότητας του Συμβουλίου. Βεβαίως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει τις πιέσεις. Ως προς την έκθεση αναχώρα, συμφωνώ με τον κύριο Ροζάτη ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πο, ε, πολλά θέματα διαφάνειας είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η, πλήττεται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, γιατί πολλές επιχειρήσεις μπορεί να μεταφερθούν ε, αλλού. Υπάρχουν πολυεθνικές οι οποίες θα πληγούν ε, αλλά το ζήτημα είναι φτάνουν το κατόφλι των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό έχει σημασία για την οδηγία, δηλαδή το ποσό που καλύπτεται ή επιχειρήσεις που καλύπτονται, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να εντάσσονται αυτές οι πολυεθνικές σε αυτή την οδηγία για να υπάρχει δικαιοσύνη με τις ε, μικρές θηγατρικές και ο συνάδελφος Κοφόντ είπε κάτι πολύ σημαντικό. Κατά την προηγούμενη συνόμια Επιτροπή ΤΑΞ μιλήσαμε για νομικά κενά. Γιατί η κυρία Ζολή αναφέρθηκε για ένα σύστημα τύπου IKEA. Κάτι τέτοιο στο παρελθόν ήταν αδιανόητο. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρόκειται για μια αγορά που είναι ανταγωνιστική, δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων και δεν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ε, ένα καθεστώς ε, μη συμβατότητα σε σχέση με τα διοικητικά συμβούλια και τους πελάτες. Μόνο έτσι θα φτάναμε σε μια πραγματική πρόοδο. Ο Επίτροπος έχει το λόγο για να απαντήσει. Καταρχήν, ως προς τη ε, θέση του Συμβουλίου. Δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξο, αλλά πιστεύω ότι η Λουξεμβουριανή Προεδρία ήταν μια καλή Προεδρία γιατί κατάφερε να ε, ε, ξεπεράσουμε σοβαρά θέματα και έφτασε και στην οδηγία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με βάση τα tax rulings. Άρα αυτό που μας ενδιέφερε ήταν η συνολική ισορροπία που επετεύχθη με αυτή την οδηγία, την οποία προέβαλε η Προεδρία του Λουξεμβούργου. Υπάρχει και πολιτική θέληση από την Ολλανδική Προεδρία να προωθήσει το πακέτο που υπέβαλα σήμερα. Βεβαίως ε, δεν προτρέχω, ούτε θέλω να προτρέξω γιατί στο Συμβούλιο υπάρχει η τάση να διαχωρίσουμε το πακέτο, δηλαδή ε, ως προς τα BEPS ε και τις άλλες πτυχές. Αυτό που θέλουμε όμως είναι μια συνολική προσέγγιση. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα διαγραμματίσει το ρόλο που πρέπει για να καθοδηγήσει το Συμβούλιο. Πρόκειται για κάτι το οποίο ε, δεν έχει προηγούμενο. Γιατί ε, εισακούεστε. Υπάρχει πίεση της κοινή γνώμης που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ως μοχλό. Σε σχέση με την τελευταία σας υπόδειξη δεν μπορώ να εκφραστώ προσωπικά γιατί είμαι επίτροπος. Ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν χαρτοφυλάκια συναδέλφων. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν παίρνω θέση επί της ουσίας σε σχέση με την υπόδειξή σας. Πρόκειται για ένα θέμα που μας απασχολεί γενικότερα η σύγκρουση συμφερόντων, κάτι το οποίο θα εμβαθύνουμε για να υπάρχει και φορολογική διαφάνεια. Δεν έχουμε κερδίσει, χρειαζόμαστε μεν τους δε, αλλά ας μην βάλουμε στο στόχαστρο το Συμβούλιο ακόμα. Μπεν Λουκέ. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ που ήρθατε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η... το όραμά σας για τις εκθέσεις αναχώρα. Είπατε ότι στην αρχή, στην παρούσα φάση, θέλετε να εισαγάγετε μια προσεκτική ε, εκδοχή το, της έκθεσης αναχώρα και να μην την δημοσιεύσετε και να αφορά αυτό τις επιχειρήσεις με ε, κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατομμύρια. Γιατί αυτός ο περιορισμό ρωτώ. Γιατί διαχωρίζονται τις ε, επιχειρήσει που έχουν λιγότερο ή περισσότερο από 750 εκατομμύρια κύκλο εργασιών. Αυτή είναι η αντίληψή σας για τις ε, ίσους όρους ε, ανταγωνισμού. Μήπως το γεγονός ότι υπάρχει και θα υπάρχει αυτό το όριο αυτό πλέον για τις επιχειρήσεις που είναι πάνω από το όριο αυτό. Οδηγήσει σε αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων όπου ενδεχομένω να δημιουργηθούν ε, θηγατρικές ε, φαινομενικά ανεξάρτητες εταιρείε προκειμένου να μην συμπεριληφθούν στις εκθέσεις αναχώρα. Και θα ήθελα επίσης να γνωρίζω το εξής μήπως θα γίνει και θα πρέπει να γίνει μία εξίσωση των επιχειρήσεων και μήπως οι μικρομεσές ε, αυτές επιχειρήσεις που πληρώνουν όπως ε, είπατε τώρα 30% παραπάνω φόρο και τελικά οδηγήσουν σε διαφορετική ρύθμιση για να διαμορφωθούν σε μεγαλύτερους ομίλους. Σε ό,τι αφορά το πακέτο σας επίσης για την ε, αποφυγή της φοροαποφυγής, έχετε κάνει ε, τέτοιες διακρίσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Θα υπάρχουν δηλαδή και σε άλλα τμήματα του πακέτου αυτού οι ε, και ρυθμίσεις για τις μικρές επιχειρήσεις. Ο κύριος Επιτρόπος. Δεν θα ήθελα να επανέλθω ε, γιατί το σκεπτικό ε, της έκθεσης αναχώρα. Πρόκειται για μια διαδικασία ε, η οποία είναι λιγότερο δαπανηρή από μια εθνική προσέγγιση και υπάρχει και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Με αυτό το ε, reporting υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο δήλωσης από το να γίνει ανακράτος. Δηλαδή υπάρχει μία συντονισμένη προσέγγιση αντιμετώπισης της φοροαποφυγής. Μιλήσαμε για τα 750 εκατομμύρια αυτό τον κύκλο εργασιών. Αυτό είναι το επίπεδο που ορίζει και ο ΩΣΑ. Αυτό είναι το κατόφλι. Άρα συμβαδίζουμε με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ. Ο κύριος Μορέλ μίλησε για τον ε, κύκλο εργασιών, το συνολικό κύκλο εργασιών σε σχέση με τον αριθμό απασχολούμενο Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχουν οι οικονομικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με το forum shopping. Και δεν μπορούμε να πούμε ως Επιτροπή τι θα κάνουν στη συνέχεια. Εάν υπάρχει λιγότερη φοροαποφυγή και λιγότερο, λιγότερο επιθετική πολιτική, τότε τα κράτη-μέλη θα είναι αυτά τα οποία θα μπορέσουν να μειώσουν το εταιρικό φόρο και έτσι να προσδώσουν ένα νέο δυναμισμό στις ΜΜΕ. Τέλος, ως προς το τρίτο ερώτημά σας, η, στην οδηγία για τη βελτιστοποίηση δεν διαφοροποιούμε αναμέγεθος επιχειρήσεων. Υπάρχει Υπάρχουν ε, ε, σχήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούν οι ε, ΜΜΕ διότι είναι δαπανηρά. Και οι επιχειρήσεις που έχουν ε, μεγάλες υπηρεσίες και μια νομική ε, πλαισίωση έχουν περισσότερες ε, διευκολύνσεις. Αλλά δεν θέλαμε να προβούμε σε μια, την, σε, μια τέτοια διαφοροποίηση στην εθνική προσέγγιση, δηλαδή στην έκθεση country by country. Με συγχωρείτε που επεκτείνουμε. Έχετε μία οδηγία αφορά την καταπολέμηση της φοραποφυγής και μία άλλη οδηγία για το CBCR. Δύο είναι οι οδηγίες. Τον Βαντερ Κάντελαρ. Ευχαριστώ, Επιτροπέ, που είσαστε εδώ πέρα μαζί μα. Θα ήθελα να σα θέσω μια ερώτηση για τον φόρο επί των χρηματοστηρικών συναλλαγών. Ε, Αναφέρθηκαν στο προσχέδιο του Δεκεμβρίου ε, κάποιες, ε, κάποια βασικά στοιχεία για τον φόρο αυτό. Και τώρα θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις μετοχές και τα παραγωγά, υπάρχει και μία τρίτη παράγραφος με άλλα στοιχεία, η οποία λέει ότι τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι για μία ανάλυση για την πραγματική οικονομία και για τα συνταξιωτικά ε, συστήματα θα πρέπει να γίνει ανάλυση και θα πρέπει να ε, ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικό αντίκτυπο και χρειάζεται και ερευνά του φορολογική βάση κάθε χώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να δοθεί μια απάντηση στην ανησυχία αυτή για τι χώρε ε, που συμμετέχουν, αλλά και για να συμμετέχουν οι χώρε που δεν συμμετέχουν ήδη για τον φόρο αυτό. Ερωτώ λοιπόν, θα μπορούσατε να μα πείτε κατά πόσον η τρίτη παράγραφο αυτή είναι εξίσου σημαντική με τι δύο πρώτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα εστιαστεί στι ανησυχίε που εκφράζονται στην παράγραφο αυτή και ίσω θα μπορούσατε να μα πείτε σήμερα ήδη πώ σκοπεύετε να το πράξετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριος Επίτροπο, λέει ο Πρόεδρο. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό και αποφασιστική σημασία μάλιστα το ότι τα κράτη-μέλη πριν της το τοποθετήθηκαν υπέρ μιας αρχής για τη φορολογία, το Βέλγιο, με τον Βέλγο Υπουργό των Οικονομικών, πρώτο-πρώτο μάλιστα, και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει το Βέλγιο έναν φόρο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το θέμα δεν είναι να παρουσιάσει η Επιτροπή τώρα πρόταση. Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή έχει πιο τεχνικό και πολιτικό ρόλο να διαδραματίσει ο πρόεδρος Γιουνκέρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε πως υποστηρίζει ένα τέτοιο φόρο. Η Επιτροπή που για χρόνια όχι είχε παραγωνιστεί αλλά είχε μπει η ίδια στο περιθώριο λέει ότι είναι παρούσα εφόσον υπάρχει η πολιτική συμφωνία. Όταν θα είναι έτοιμο το κείμενο θα συζητηθεί με τους 28 Και παραλαμβάνω, δεν πρόκειται για κοινοτική μέθοδο τη ενισχυμένη συνεργασία. Τώρα τη λέει συμφωνία, και δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε γιατί εξορισμού το σύνολο το όλον τη συμφωνία είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Δεν θα επιλέξω εγώ κανένα κομμάτι τώρα. Αλλά με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν το Δεκέμβριο, με βάση αυτά, μας μένουν μερικοί μήνες μέχρι τα τέλη Ιουνίου για να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους του φόρου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στη συνέχεια θέματα τα οποία φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνήσετε πως δεν είναι αμεληταία το συντελεστή του φόρου και τον προορισμό του προϊόντος αυτού του φόρου. Η συμφωνία της 1ης Δεκεμβρίου πάντως είναι καθοριστική σημασίας. Δεσμεύει τα μέρη, γιατί δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν μέχρι τα τέλη, τα τέλη Ιουνίου την απόφαση αυτή και είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα εν λόγω κράτη μέλη και εμείς ως Επιτροπή προσφέρουμε ε, την τεχνογνωσία και την πολιτική υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Εγώ όπως είπα δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα να τοποθετηθώ για κάποιο σημείο συγκεκριμένο ενός κειμένου το οποίο υιοθέτησαν οι Υπουργοί. Ευχαριστώ πολύ, Σοσιαλιστές Δημοκράτες, κυρία Γκόμες. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Τα πορτογαλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, στα τέλη του 2015 δημοσίευσαν ε, κατάλογο των μεγάλων εταιριών, κυρίως πετρελαϊκών και ε, στον ενεργειακό τομέα, Φερρυπίν της Αναγκόλ, της Αγκόλας και άλλες μεγάλες τράπεζες με έδρα τη Μαδέρα που τους ωφελεί ιδιαίτερα φορολογικά λόγω των διευκολύνσεων που προσέφερε το πορτογαλικό κράτος με όφελος περί το 1 δις ευρώ συνολικά. Βέβαια, εγώ σκοπεύω να αποστείλω επιστολή στην κυρία Φερστάκερ για να την παρακαλέσω να εξετάσει αν πρόκειται για παράνομες κρατικές ενισχύσεις αλλά ερωτώ εσάς, γιατί παραμένει σιωπηλή και τυφλή η Επιτροπή σε όλα αυτά τα θέματα και κυρίως με τη δουλειά που έχουμε κάνει και εμείς από εδώ και εσείς από την πλευρά σας. Και επίσης καθώς γνωρίζουμε ότι η νομοθεσία που ενέκρινε το Συμβουλίο για την αυτόματη ανταλλαγή αποφάσεων σχετικών με τις προκατακτικές φορολογικές αποφάσεις μπορεί να μην καλύπτει τις εν λόγω συμφωνίες που αφορούν χώρες με έδρα ένα κρατος μέλος και μία τρίτη χώρα. Και όπως είπε η κυρία Φερέιρα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμένου, γιατί δεν προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαγάγει την φορολογική ισονομία εναντί του, ε, των κρατών, ώστε και ο φορολογούμενος να βλέπει ότι μπορεί να μειωθεί η φορολογία εκείνου ο οποίος είναι πιο φτωχός και ότι συλλέγεται πεστρός από εκείνον που μπορεί να πληρώσει πεστροφόρο. φόρο ο αρμόδιος δε υπουργό στην Πορτογαλία έχει δηλώσει ότι οι πιο πλούσιες οικογένειες Πορτογαλίας που θα έπρεπε να καταβάλουν 25% του φόρου από το εισόδημά τους, μόνο 0,5% καταβάλουν λόγω των φορολογικών εξαιρέσεων, ευνοϊκών μεταχειρήσεων και απαλλαγών που βέβαια χορηγούνται σε απόλυτη αδιαφάνεια. Γιατί δεν αντιδράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καταρχάς. Και για να συνεχίσουμε στη γραμμή της εκθέσεως Φερέιρα έχει στήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον, ε, ε, ε, μια ενιαία βάση υπολογισμού του φόρου για τις επιχειρήσεις, την αντιμετώπιση της μεταφοράς κέρδους, την αναθεώρηση της οδηγίας για τη royalties. Τι γίνεται για αυτά όλα κύριε Επιτροπέ. Απάντηση. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Η πρώτη για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Η απάντηση είναι ότι η αρμοδιότητα είναι τη Γενική Διευθύνσεω Ανταγωνισμού. Η κυρία Φερστάγκερ ασφαλώς θα χαρεί να λάβει την επιστολή σας. και θα σας απαντήσει. Υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο και πολύ αυστηρές προδιαγραφές για το κατά πόσο μπορούν να ιδρυθούν ελεύθερες οικονομικές ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα ήταν ένας τρόπος ε, να διευκολύνουν κάποιες περιφερειές τους στα κράτη-μέλη για να τους δώσουν περισσότερες ευκαιρίες κτλ. Και πρόκειται πέν για αρμοδιότητα των κρατών μελών των ίδιων, αλλά αυτό αφορά επιχειρήσεις που έχουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην ελεύθερη οικονομική ζώνη και δεν μπορεί αυτό να ε, αποβαίνει ει βάρο της λειτουργίας άλλων αντίστοιχων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη οικονομική ζώνη, σημειώνω, δεν είναι ζώνη εκτός του νόμου, άρα ισχύουν όλες οι διατάξεις νομοθετικές και βέβαια και αυτό το σχετικό με τη διάταξη και σχετικά με τις εκθέσει ανακράτο. Ε, οι προτάσει μας θα ισχύσουν και για τη Μαδέρα όταν έρθει όλα βεβαίω και και στη συνέχεια της εκθέσεως Φερέρα Τόιρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει οι διατάξεις κατά των καταχρήσεων ε, που στόχο έχουν να αποτρέψουν ε, την κατάχρηση ευκαιριών από επιχειρήσεις και την αποφυγή καταβολής φόρου. Έχουμε προτείνει λοιπόν την ενίσχυση αυτών των διατάξεων και την προσαρμογή στο ταχύτερο δυνατό ε, των προτάσεων για την οδηγία Μέρφη και αντίστοιχα και την οδηγία για τις συγχωνεύσεις και για τα ε, για τους τόκους από προσαρμοσμένα έσοδα. Ευχαριστώ πάντως για την ερώτηση. Και τώρα ο κυρίος Ενρικέ Καλβέτσον, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτό το πακέτο που υποβάλατε, που είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής των μικρών βημάτων για την οικοδόμηση Ευρώπης που πλέον δεν αρκεί. Είμαι ο τελευταίος ομιλητής και θα ήθελα να σας υποβάλω τέσσερις ερωτήσεις, άμεσες ερωτήσεις. Είπατε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από τον όσα. Γιατί δεν μιλάμε για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γιατί δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Ίσως θα έπρεπε. Μιλήσαμε για το Λίχτενστάιν, ίσως και την Ελβετία και το ε, Μονακό. Μπορείτε να λάβετε υπόψη και το Γιβραλτάρ, υπάρχουν ε, και άλλοι φορολογική παράδεισοι. Έχετε κάτι να πείτε για αυτούς. Εδώ μιλάμε για αυτό το τείχος χρήματος που ολοένα και ορθώνεται έναντι των ε, ψηφοφόρων μας. Ως προς την φοροαποφυγή δεν θα ήταν σκόπιμο αντί να ακολουθούμε μία ειδική νομοθετική διαδικασία, νομική διαδικασία διαβούλευσης, να είμαστε από κοινού νομοθέτης και εμείς μαζί με το Συμβούλιο. Ακόμα και αν αποχώρησε η κυρία Ζουλή, θα ήθελα να πω ότι ακούω στην ΕΟΚΕ να γίνεται λόγος εδώ και 20 χρόνια για το θέμα της φορολογικής βάσης. Μέχρι πότε θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα χάσματα που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ειλικρινία σας η οποία δίνει μία ζωντάνια στη συζήτηση και βοηθάει συνάμα ως προς τις ε, σχέσεις ε, με τον Όσα. Εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι προς την ίδια κατεύθυνση με τον Όσα για, τη, για την ιστορική αγορά. Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είπα ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου. Γίνονται συζητήσεις τεχνικού τύπου και θα βρούμε παγκόσμιες λύσεις. Δεν είναι μικρά τα βήματα, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, αλλά δεν είναι το τελευταίο. Τα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα θα αντιμετωπιστούν με την ώρα τους. Ως προς εσωτερικούς φορολογικούς παραδείσους δεν χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία. Δεν υπάρχουν εσωτερικοί παράτηση. Υπάρχουν χώρες που έχουν άλλη φορολογική βάση, πιο πλεονεκτική. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν τις απαλλάσσουμε. Το είπα και για την Ιρλανδία. Δεν θα επανέλθουμε στο 12%. Δεχόμαστε την εθνική κυριαρχία, αλλά δημιουργούμε ένα πλαίσιο <coughs> λειτουργίας έχουμε κάνει τις συμφωνίες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται, γίνεται άρση ε, απορρίτου στην Ελβετία, στο Λίχτενστάιν, στην Ανδόρα και στο Σαν Μαρίνο και στο Μονακό την επόμενη εβδομάδα. Άρα έχει αρθεί, έχει πεθάνει το τραπεζικό απόρριτο στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια γιγάντικα, γιγάντια εργασία που πραγματικά έγινε. Δέχομαι ε, αυτά που είπατε για το ρόλο του κοινοπούλου. Υπάρχουν όμως οι συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να τηρήσουμε. Το τελευταίο θέμα είναι μεγάλη σημασία, ύψιστη της σημασίας, η φορολογική βάση. Δυστυχώς για την οδηγία φορολογικής βάσης δεν υπήρξε συμφωνία στο Συμβούλιο. Θα την ξαναπροωθήσουμε. Η φορολογική βάση είναι ένα σκόπιμο μέσο για να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή. Θα ε, δεχτούμε τα προνόμια που έχουν ορισμένα κράτη-μέλη, Άλλα κράτη θέλουν εναρμόνιση, φορολογική εναρμόνιση, αλλά όχι. Αυτό το δεχόμαστε. Αλλά ο εταιρικός φόρος δεν είναι το βασικό κριτήριο για τη μεταφορά κερδών. Θα πρέπει όμως να προωθήσουμε μακροχρόνια την ε, φορολογική βάση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτό το θέμα της ενιαίας φορολογικής βάσης εντάσσεται στα μικρά βήματα τα οποία θα κάνουμε. Και φυσικά θα επανέλθουμε και θα επανέλθω και εγώ εδώ ενώπιον σας ε, για να μιλήσω για ένα νέο ε, σχέδιο φορολογικής βάσης. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε πίτροπε, ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την ζωντανή και πλούσια ανταλλαγή απόψε. Μπορέσαμε να συνεργαστούμε στενά προς την ίδια κατεύθυνση και θα προσπαθήσουμε να πιέζουμε πολιτικά αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η πολιτισμική βάση, η βάση σκέψης, δηλαδή από τον αθέμητο χαρακτήρα του ανταγωνισμού και της φορολογικής βάσης θα φτάσουμε σε μία πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα. Πέρσι, όπως γνωρίζετε, καταφέραμε να έχουμε ε, την άρση του τραπεζικού απορρίτου, τώρα αποφανθήκαμε και για τα tax rulings, άρα πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μια συμφωνία με βάση τις συστάσεις του όσα και μετά την πλήρη εναρμόνιση του, της ε, εταιρικής φορολόγησης. Η Επιτροπή Τάξ θα ακούσει και τους επιτρόπους Φερστάγκερ και Χίλ και σας υπενθυμίζω ότι την ε, Δευτέρα ε, στις 18.30 θα συνέλθουν οι συντονιστές και στις 29 στις 15.30 θα ακούσουμε την Ολλανδική Προεδρία που ελπίζω να μας επιβεβαιώσει τις προθέσεις σας. Θέλετε κάτι να πείτε? Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τους συναδέλφους για την άκρο ενδιαφέρουσα συζήτηση που δείχνει ότι ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βοηθήσει να εισακουστούν και να υλοποιηθούν αυτές οι, προτάσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ ε, κύριε Επίτροπε, με τη σειρά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Λύεται συνεδρίαση.